Chers collègues, si vous voulez bien prendre καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Η ημερήσια διάταξη σας έχει διανεμηθεί. Δεν έχω λάβει κάποια ιδιαίτερα σχόλια. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίθηκε. Με μόνη διαφορά ότι στο σημείο 3 επρόκειτο να ψηφίσουμε για το κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Το αίτημα αφορά το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Είναι μια βελγική και ιρλανδική υπόθεση και η ομάδα εργασίας μας δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Ζητήσαμε από την Επιτροπή Προϋπολογισμού να μας πει αν μπορούσαμε να αποσυνδέσουμε τις δύο περιπτώσεις και να τις εξετάσουμε με διαφορετικό τρόπο, διότι στην περίπτωση της Ιρλανδίας Μιλάμε για τη συνέχεια της επιπτώσεις ε, της, ε, των απολύσεων στην επιχείρηση Dell μετά από πρόταση της ομάδας εργασίας απευθυνθήκαμε στους επιτρόπους Κρούς και Σπίτλε για να μας δώσουν διευκρινήσεις για το αποτελέσμα της εξέτασης για το θέμα αυτό της Επιτροπής. Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Μέχρι τώρα δεν έχουμε την απάντησή του για να ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις. Γι' αυτό σας προτείνω να αναβάλουμε την εξέταση και την ψηφοφορία αυτών των γνωμοδοτήσεων ε, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση μας ε, Για το 2 υπάρχει, να σας πω ότι υπάρχει web streaming των εργασιών μας που μπορεί και να τις παρακολουθείς απευθείας στο διαδίκτυο και έχουμε μία αίθουσα στο 1G2 όπου όσοι δεν χωράνε εδώ μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες μας και ελπίζω ότι το σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα από την τελευταία φορά. Θέμα 4 στην ειδήσια διάταξη. Αυτός, ε, αυτό θα είναι και το κυρίως θέμα μας για σήμερα, εφόσον θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων για δύο μελέτες, 4α και 4β, τις οποίες προτείνω να εξετάσουμε τη μία μετά την άλλη, διότι δεν πρόκειται ακριβώς για τους ίδιους ομιλητές, οι συνομιλητές, ξεκινώντας με τη μελέτη η οποία έγινε από το Labor Associates SLA για τις προκλήσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η μελέτη αυτή, η οποία ανατέθηκε από τους προκατόχους μας, θα είναι τελικά διαθέσιμη από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο τέλος Οκτωβρίου αλλά τα βασικά της σημεία, τα κυριότερα σημεία της υπάρχουν ήδη στο τραπέζι τα έχουμε μπροστά μας και όταν θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με του αρμόδιους ε, επιτρόπους και την μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο ήδη από σήμερα να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για να ενημερωθούμε. Θα γίνει πρώτα μια παρουσίαση της ίδιας της μελέτης και ευχαριστώ τον κύριο Ρικάρντο Ροντρίγκε της εταιρεία που ανέλαβε την διεξαγωγή της μελέτης για το γεγονός ότι μας την παρουσιάσει και μετά θα δώσουμε το λόγο στους κοινωνικούς εταίρους για να αντιδράσουν και να, δούμε τις δικές τους αντιδράσεις και να μας πούν τι πιστεύουν για αυτή τη μελέτη. Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Ροντρίγκο Ροντρίγκες, Νομίζω ότι ο κύριος Higgins, νομίζω, θέλει να πάρει το λόγο. Πρόκειται για διαδικαστικό, κύριε Higgins. Χωρίς μικρόφωνο. Σχετικά με την πρότασή σας να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Για το σημείο 3 προτείνατε να αναβληθεί η εξέταση αυτού του θέματος. Συμφωνώ με την πρότασή σας, αλλά θα μπορούσαμε στις συζητήσεις, να, να, να συμπεριλάβετε στις συζητήσεις την παράδοξη θέση της Επιτροπής η οποία έδωσε στην Dell Corporation 40 εκατομμύρια για να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας στην Ιρλανδία με θέσεις εργασίας στην Πολωνία. Και ποιο είναι ο στόχος ποιος θα είναι ο σκοπός μιας τέτοιας στρατηγικής γιατί ακριβώς πρόκειται. Δεν θέλω να βρεθούν αντιμέτωποι μεταξύ τους οι εργαζόμενοι στις δύο αυτές χώρες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθούμε σχετικά. Μα γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα ψηφίσουμε σήμερα για το βελγικό αίτημα. Ε, λάβαμε σε μια πρώτη φάση το αίτημα του Βελγίου το βελγικό αίτημα κατόπιν συμπληρώθηκε με ένα ταυτόχρονο παράλληλο αίτημα της περίπτωσης της Ιρλανδίας, της υπόθεσης της Ιρλανδίας, που αφορά την εταιρεία Dell, όπως σας είπα και είπατε κι εσείς. Ακριβώς λοιπόν για αυτά που μας είπατε, πρότεινα στην ομάδα εργασία, η οποία δέχθηκε, να αποσυνδέσουμε τι δύο περιπτώσει, Διότι τόσο στη βελγική περίπτωση αντιμετωπίζουμε μια αρκετά κλασική περίπτωση αιτήματο κινητοποίησης του Ταμείου και ε, όπως θα δούμε όταν εξετάσουμε σε βάθος το θέμα, έχουμε τη σωστή ε, ε, αντιμετώπιση από όλους τους ενδιαφερόμενους, ενώ αντίθετα στην Ιρλανδική περίπτωση τα πράγματα είναι τελείως παράλογα. Η κατάσταση είναι τελείως παράλογη. παράλογη. Διότι στην, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μία, η μία διεύθυνση κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από κάποια άλλη διεύθυνση, δεν υπάρχει σύμπνοια στο σώμα Υπάρχουν αντιθέσεις, έχουμε αντα... Ε, θέσεις σε ανταγωνιστική ε, υπόθαλψη ανταγωνισμού ανάμεσα ε, στους εργαζόμενους δύο διαφορετικών χωρών. Ο σκοπό όμω είναι να διατηρούμε τι θέσει εργασία εκεί όπου υπάρχουν, όχι να τι μεταφέρουμε αλλού. Δεν θα μπούμε στο βάθο αυτού του θέματο, επειδή είπαμε ότι θα το αναβάλουμε αλλά οι ανησυχίες που διατυπώσατε ανταποκρίνονται, συμφωνούν απόλυτα με εκείνες που διατύπωσαν τα μέλη της ομάδας εργασίας. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να αναβάλουμε τη συζήτηση για όλο το θέμα. Γράψαμε στους δύο αρμόδιους επιτρόπους, κινητοποίησαμε την Επιτροπή Προϋπολογισμού όταν θα εξετάσουμε το ε, Ιρλανδικό αίτημα σχετικά με την εταιρεία Dell θα μπορέσουμε, ελπίζουμε, να πάρουμε μια απόφαση που δεν θα αντιβαίνει τα συμφέροντα της εταιρείας Dell, αλλά έχοντας προηγουμένως, έχοντας προηγουμένως διευκρινίσει όλα αυτά τα θέματα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να αρχίσουμε να έχουμε τώρα μια συζήτηση, επειδή, όπως σας είπα, όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες μας, αυτή η συζήτηση έχει αναβληθεί. Επειδή όμως μου ζητάτε το λόγο, θα σας τον δώσω βεβαίως, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομος. Κύριε Ντερόζα. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που άργησα λίγο. Η μόνη ε, ανησυχία μου είναι ότι κάνουμε σήμερα να μην καθυστερήσει ε, την έκβαση της υπόθεσης για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους. Ο πρόεδρος μπερόσο επισκέφθηκε την Ιρλανδία και είπε ότι θα υπάρξει ε, απάντηση, θα ήταν καταστροφικό για τους εργαζόμενους και για την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν ό,τι κάνουμε καθυστερήσει την ε, χρηματοδότηση για τους εργαζόμενους αυτούς. Ε, Συμφωνώ απόλυτα και συμμερίζομαι απόλυτα την ανησυχία σας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής όμως, όταν πήγε στις 19 Σεπτεμβρίου στην Ιρλανδία, δεν τήρησε τις σωστές διαδικασίες. Δεν μπορούσε να υποσχεθεί κάτι που δεν είχε ακόμα επικυρωθεί. Ήταν απλά μια πρόταση της Επιτροπής που έπρεπε κατόπιν να επικυρωθεί από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχή, κάτι που δεν συνέβη, αρχές, κάτι που δεν συνέβη. Αλλά αντιλαμβάνομαι αυτά που μας λέτε, ότι δεν πρέπει να θυγούν τα συμφέροντα των εργαζομένων στην Ιρλανδία. Και γι' αυτό θα εξετάσουμε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν μπορούμε για αυτού τους λόγους να γνωρίσουμε όλες τις ασυνέπειες της διαδικασίας που εφαρμόστηκε μέχρι στιγμή και τη μη τήρηση των διαδικασιών. Κάτι που ισχύει και για την συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι συμμεριζόμαστε απολύτως και εμείς τις ανησυχίες σας. Ας επανέλθουμε λοιπόν τώρα στο θέμα 4. Ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή μας και τους προσκεκλημένους μας που έκαναν λίγη υπομονή, αλλά ήταν σημαντικό να διευκρινιστεί αυτό το σημείο, το θέμα που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Ρικάρντο Ροντρίγκε, ο οποίος σε 15 περίπου λεπτά ελπίζω θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήγαγε για την στρατηγική της Λισαβόνας 2000-2010. Κύριε Ροντρίγκες, έχετε το λόγο. Merci, merci, Σας ευχαριστώ πολύ. 15 λεπτά για να σας συνοψίσω μία δεκαετή εργασία είναι πολύ λίγος χρόνος. Ε, θα χρησιμοποιήσω αυτά τα λεπτά και θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω τα τεκτενόμενα κατά τηλεγραφικό τρόπο. Για να μην γίνει ε, παρανόηση του νοήματος αυτής της εργασίας. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι η μελέτη αυτή αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας ως προς την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Αυτή την εντολή είχαμε λάβει και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η στρατηγική της Λισαβόνας, κάτι το οποίο είναι μια επίπονη εργασία και πολλές φορές ε, ειδικά το δεύτερο τμήμα, είναι δύσκολο. Δηλαδή, ε, όπως εξελίσσεται μετά το 2005. Το πρώτο τμήμα ε, είναι το σκεπτικό αυτής της ε, στρατηγικής 2000-2005. Δεύτερον, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ποιοτικών και ποσοτικών. Και τρίτον, θα ανταποκριθούμε σε ορισμένα στοιχεία, επιμέρους στοιχεία και υποδείξεις για το μέλλον, μετά το 2010 δηλαδή. Να σας υπενθυμίσω πώς έχει η στρατηγική της Λισαβόνας, δηλαδή γεννήθηκε το 2000 για την στρατηγική της απασχόλησης έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη ένα la agenda... και η ατζέντα της Λισαβόνας είναι μια στρατηγική αναθεώρησης μακροχρόνια και αυτό αποτελεί ένα σύνολο πολιτικών φιλοδοξιών που βασίζονται στα κράτη-μέλη, στη θέλησή τους. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αναλαμβάνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και σε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες, δηλαδή στον τομέα της απασχόλησης. Γι' αυτό θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε ορισμένα συστήματα όπως την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Θα θυμόσαστε ότι το βασικό μας γνωμικό ήταν να αντιμετωπίσουμε την ε, οικονομία υπό μία πιο δυναμική θεώρηση, με μία μεταρρυθμιστική ατζέντα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, αναλύσουμε και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία που είναι οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές μας στο παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, Πέρα από την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού θα πρέπει να ορίσουμε και ποσοτικούς στόχους, targets που γνωρίζετε και στους περισσότερους επήλθε μία, ένα συμβιβασμό για το 2010 σε σχέση με ένα 10% απασχόλησης όπου ένα 50% να αφορά και γυναίκες και επίσης να υπάρχει ένας απότερος στόχος μέχρι το 2050. Όλα αυτά είναι καινοτόμα στοιχεία και αποτελούν στοιχείο ενός πολύ σοβαρού συμβασμού και δέσμευσης. Θα πρέπει να τονίσω ότι επήλθαν πολλές αλλαγές στη στρατηγική της Λισαβόνας διαχρονικά με μία ανελικτική δυναμική πορεία όπου μπορούμε να δούμε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η εκκίνηση μέχρι το 2003, όπου στον τομέα της απασχόλησης είχαμε τέσσερους ε, κοινούς στόχους, δηλαδή τέσσερις πυλώνες που γνωρίζετε πολύ καλά η προσαρμοστικότητα, η ισότητα ε, ευκαιριών, η εξελιξιμότητα και επίσης και το τέταρτο, ο τέταρτος πυλώνας που είναι το περιβάλλον, όπως όρισε το Γκέτεμπορκ. Το 2003 έγινε μία αλλαγή η οποία συμβαδίζει, συμβάδιζε με τους γενικότερους στόχους, τουλάχιστον στη διατύπωση τηλεγραφικά θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή ε, όρισε το 2003 ως απότερο στόχο την πλήρη απασχόληση και την συμπερίληψη στην αγορά εργασίας τους βασικούς στόχους. Επίσης άλλαξε το σύστημα με τους 10 συμβιβασμούς για την περίοδο 2003-2005. Μέχρι το 2005 λοιπόν ε, την κατανομάζουν αυτήν την περίοδο Λισαβόνα 1 η ακαδημαϊκή. Στη συνέχεια έγινε μία κριτική ε, σκέψη και περισυλλογή από έμπειρογνώμονες υψηλού επίπεδου και με βάση τη στρατηγική του 2002 για την στρατηγική της πλήρης, της πλήρους απασχόλησης θεωρήθηκε λοιπόν ότι δεν λειτουργεί επαρκώς η στρατηγική της Λισαβόνας. Υπήρχαν προβλήματα συντονισμού καθώς και ορισμού ποσοτικών στόχων και θεωρήθηκε ότι ορίσαμε πληθώρα στόχων που δεν είναι αποσαφηνισμένοι Άρα το 2005 αυτό το επίπεδο, αυτή η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου όρισε την στρατηγική από το 2005 και μετά και αλλάζει βεβαίως ε, ο στρατηγικός ε, στόχος, η απότερη στρατηγική στόχη. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το 2004-2005 ε, είχαμε και τη διεύρυνση με τα νέα κράτη-μέλη, το οποίο ήταν ύψης της σημασίας. Και είχαμε και τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 που εκκίνησε αυτή τη νέα στρατηγική της Λισαβόνας που γνωρίζουμε σήμερα με ορισμένα ανελικτικά στοιχεία, εξελικτικά στοιχεία. Το πιο βασικό σημείο αυτής της αναθεώρησης είναι τα εθνικά σχέδια μεταρρύθμισης όπως τα όρισαν τα κράτη-μέλη και όπως τα κοινοποιούσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχολησιμότητα που να εντάσσονται σε μάκρο και μικρο οικονομικούς στόχους έτσι ώστε να έχουμε δύο κύκλους 2005-2007 ανά τρία χρόνια και τώρα βρισκόμαστε στο τέλος του δεύτερου κύκλου. Αυτή ήταν η βασική διάρθρωση που γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και θα πρέπει βεβαίως να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα. Καταρχήν, τι έγινε με τους ποσοτικούς στόχους, πώς εξελίχθηκαν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, βεβαίως υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοί στόχοι, αλλά δεν έχω χρόνο να επεκταθώ σε αυτούς. Μία ανάλυση των διαρθρωτικών δικτών που χρησιμοποιούνται στο, για το σύνολο των ποσοτικών στόχων μας οδήγησαν σε ορισμένα συμπεράσματα. Καταρχήν, μέχρι το 2007-2008 έχουμε στοιχεία τα οποία είναι εξελικτικά, εξελικτικής φύσης για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης για να δούμε και τις τρευλώσεις επέρχονται στην αγορά. Και βεβαίως αυτή η στρέβλωση θα συνεχιστεί και το 2010. Αυτό θα πρέπει όμως να το δούμε πολύ προσεκτικά αυτά τα, αυτές τις ε, προκαταρκτικές σκέψεις και το 2010 θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση σε σχέση με τους στόχους του 70% του δίκτυα απασχολησιμότητας, τα κάτι το οποίο μας ε, ε, οδηγεί στο ότι βρισκόμαστε στο 65% μέχρι το 2008. Υπάρχουν όμως χώρες, όπως οι βόρειες χώρες, ε, Φιλανδία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκονται κάτω από αυτό το, το στοιχείο. Αλλά μέχρι το 2008 φτάσαμε σε αυτούς τους ε, στόχους. Τις έφτασαν, ε, τους έφτασαν αυτούς τους στόχους αρκετές χώρες. Υπάρχουν ε, χώρες που βρίσκονται πολύ κοντά, η Σλοβενία, οι Βαλτικές χώρες και άλλα κράτη τα οποία βεβαίως είχαν χειρότερες επιδόσεις. Το συνολικό αποτέλεσμα, δηλαδή ο μέσος όρος μας οδηγεί σε ένα έλλειμμα πέντε μονάδων κάτω από το προβλεπόμενο. Καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα ως προς την συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά παρά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και πολλές χώρες ε, υπερέβησαν το 70% ενώ άλλες ε, προώθησαν τα τελευταία 8-9 χρόνια αρκετά σημεία σε σχέση με τη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Δηλαδή ε, έχουμε ένα 59% μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρίτος δείκτης, ο οποίος είναι εμβληματικού χαρακτήρα, αφορά την συμμετοχή στην αγορά εργασίας εργαζομένων άνω των 55. Και εδώ είχαμε πολλές εξελίξεις όπου πολλές φορές λειτουργήσε καλά το όλο πλαίσιο. Άλλοι όμως βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό το στόχο του 50%. Βρισκόμαστε σε ένα 45%. Θα ήθελα να ε, κοινοποιήσω και ένα-δύο ακόμα στοιχεία, αλλά ενδεχομένως υπάρξουν και ανακύψουν και ερωτήσεις μετά από την παρουσίαση. Τα αποτελέσματα είναι άνισα σε χώρες που έχουν ε, προβλήματα να φτάσουν σε αυτούς τους ε, ποσοτικούς στόχους και στον κοινωνικό τομέα αντιμετωπίζουμε προβλήματα γιατί πολλές φορές παιδιά εγκαταλείπουν, ναι, εγκαταλείπουν το σχολείο και γι' αυτό ανακύπτουν πολλές ανισότητες. Αυτές οι ανισότητες εντάσσονται σε, διάφορες, σε διαφοροποίησεις κατά τα έτη 2004-2007 με πολλές απώλειες και είχαμε να κάνουμε και με άτυπες συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν με τους ε, εργαζομένους. Επίσης, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ε, πρόσκομα ως προς την ε, στρατηγική της Λισαβόνας, διότι υπάρχουν μεταβλητές που δεν μπορούμε να απομονώσουμε εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, η στρατηγική Τη στρατηγική της Λισαβόνας δεν μπορούμε να την κρίνουμε μόνο ποσοτικά. Υπάρχουν ε, θέματα τα οποία σχετίζονται γενικότερα με, την, ε, με το πώς εντάσσονται μακρόπνοα στη στρατηγική της Λισαβόνας. Και αυτό που έχει σημασία είναι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού στον τομέα της απασχολησιμότητας και στο τομέα της ε, κοινωνικής συμμετοχής. Έγιναν πολλές κατά περίπτωση ε, μελέτες με θετικά αποτελέσματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη κατανόηση από τα κράτη-μέλη. Γιατί πολλές φορές σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο ένα κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα πρέπει να υπάρχει και μία κοινή θεώρηση ως προς τις ε, μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να προωθήσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι τακτικές περί είναι εθνικού χαρακτήρα. Και αυτό που έχει σημασία είναι η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών απασχολησιμότητας στα κράτη-μέλη η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, μάλλον με αυτή την ε, θετική αναγνώριση, καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν μελετηθεί πολύ περισσότερο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με καινοτόμα στοιχεία με βάση αυτή τα κοινά στοιχεία συντονισμού. Και αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα αξιοποιήσουμε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως προς την ε, κοινωνική προστασία και την ε, ένταξη στην αγορά εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μία ιδιαίτερη μελέτη στην οποία δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Λισαβόνας βασίζεται στα κράτη-μέλη και δεν βασίζεται μόνο στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει ένα κοινοτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με τις ε, ευρωπαϊκές προσπάθειες έτσι ώστε να μπορούν να παγιωθούν ε, ορισμένες δυνάμεις εργασίας ε, μέσα στα πλαίσια της έγκρισης οδηγιών, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως η χρηματοδότηση και τα, οι τελευταίες ε, δημοσιονομικές προβλέψεις 2007-2013 που εντάσσουν σε αυτό το υπερεθνικό πρόγραμμα που αποτελούν μια παράλληλη οδό εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που εφαρμόζουν την στρατηγική καθεαυτή και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινοτικό προπολογισμό για την στρατηγική αυτή. Και τα δημοσιονομικά βασίζονται στα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να προβούν σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων. Άρα το χρηματο, τα χρηματοδοτικά μέσα όπως το Ταμείο Σύνοχης και το Κοινωνικό Ταμείο ενισχύονται και σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πριν από το 2007, πριν από την έγκριση των ε, τελευταίων δημοσιονομικών ε, πρόπτικων ε, επήλθαν πολλές αλλαγές και τώρα και τα δύο αυτά ταμεία μέσω του, των κανονισμών του συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Υπάρχουν και άλλα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης που εντάσσεται στη στρατηγική της Λισαβόνας. Κατά τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να δούμε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας στις εθνικές πολιτικές απασχολησιμότητας. Δηλαδή, οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές, τι επιπτώσεις είχαν. Τα τελευταία 8 με 9 χρόνια είδαμε ότι τα κράτη-μέλη φύρμωσαν διάφορες μεταρρυθμίσεις ως προς την αγορά εργασίας. Και ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήρες γραμμές απασχόλησης. Καθίσταται σαφές ότι στις συζητήσεις με τους αξιωματούχους που ασχολούνται με τις ε, μεταρρυθμίσεις απασχολησιμότητας δεν υπάρχει αυτός ο καταλογισμός. Και οι πρόσφατες μελέτες συνδέονται άμεσα με ορισμένες από τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης που έχουν εισαχθεί στη στρατηγική της Λισαβόνας. Πέρα από αυτές τις επιπτώσεις μπορούμε να σκεφτούμε και άλλες ε, μεταρρυθμίσεις όπως στη Γερμανία και σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν στοιχεία ευελιξίας και που όλα ένα και επεκτείνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με την επίπτωση της στρατηγικής της Λισαβόνας στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης. Έχουμε να κάνουμε με δύο τρόπους ή τύπους, δηλαδή τη δημιουργία νέων στοιχείων ως προς την πολιτική απασχολησιμότητας που δεν υπήρχαν μέχρι τούτε. Ή... Ε,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 quasi oggettivamente. ένα ερώτημα αντικειμενικά, δηλαδή εάν η στρατηγική της Λισαβόνα σε μία ε, φάση δυσκολίας όπως την παρούσα ε, επιβεβαιωθεί ή χρειάζεται ορισμένε ε, μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές. Εγώ τάσομαι υπέρ της πρώτης, του πρώτου σκεπτικού. Εάν η στρατηγική της Λισαβόνας είχε εφαρμοστεί σωστά από τα κράτη-μέλη, τότε η Ευρώπη πρόσφατα δεν θα αντιμετώπιζε τόσες δυσκολίες από αυτές που αντιμετωπίζει. Βεβαίως υπήρχαν ανισότητες μεταξύ κρατών και άρα αναπόφευκτα θα έπρεπε να βρεθεί ένα σημείο εκκίνησης που δεν ήταν ισόρροπο. Όμως, όπως ε, μας επιβεβαιώνουν στοιχεία που λάβαμε, αυτό που έχει σημασία είναι η θέληση των μεμονωμένων κρατών μελών. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα άνοιγμα της ψαλίδας κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε σε επίπεδο πολιτικής θέλησης. Τι έχει σημασία για την Ευρώπη. Αυτό που έχει σημασία είναι να βγούμε από την παρούσα κρίση. Εμείς χρειαζόμαστε ένα μοντέλο ανταγωνιστικότητας το οποίο να έχει ένα σημείο επικέντρωσης. Νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι η ποιότητα των ε, στοιχείων που παράγουμε και πώς τα παράγουμε. Διότι οι συνθήκες σε άλλες, σε χώρες που μας ανταγωνίζονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αφορούν το, ποιοτικό τους προφίλ στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Εμείς δεν μπορούμε να παραμείνουμε απομονωμένοι και να μην φτάσουμε σε, αυτό το, σε αυτή τη σημαντική ημερομηνία για την επίτευξη της στρατηγικής της Λισαβόνας, προσπαθώντας να ανακτήσουμε αυτό που χάσαμε καθοδόν, αλλά μην χάσουμε την κατεύθυνσή μας. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι η ευημερία των λαών και θα πρέπει να αποτελέσει θεμέλιο του μοντέλου ανταγωνιστικότητας. Επίσης, ε, στην καινοτομία θα πρέπει να βασιζόμαστε για την εκπαίδευση, ξεκινώντας από το σχολείο έτσι ώστε να δώσουμε ταυτότητα στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και ποιότητα. Ποιότητα ως προς το χώρο εκμάθησης. Θα πρέπει να μην υπάρχει προστατευτισμός, αλλά θα πρέπει να ρυθμιστεί η αγορά για να μην έχουμε επανασύνθεση μονοπωλίων που διαβλέπουμε εδώ και εκεί. Τέλος, η στρατηγική της Λισαβόνας δεν αφορά μόνο την πολιτική σφαίρα, δηλαδή τα θεσμικά όργανα. Καθίσταται σαφές ότι χρειάζεται μία ενίσχυση μεταξύ ε, σχέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, αλλά επίσης η στρατηγική της Λισαβόνας θα κινηθεί μόνο εάν παράλληλα η σχέση μεταξύ κοινωνικών φορέων συνάδει με τους στόχους της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Μπορούμε να ανακτήσουμε πάρα πολλά σε αυτό το έδαφος, δηλαδή δεν αμφισβητούμε την αυτοδυναμία των κοινωνικών εταίρων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια έξι ισορρόπηση, διαφορετικά θα έχουν επιπρόσθετες δυσκολίες ε, τις οποίες απευχόμαστε. Η κυρία Σουέτερ και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα, πέρα από τις ε, παρατηρήσεις που θα κάνω για την στρατηγική της Λισαβόνας, ε, θα ήθελα να πω ότι η μελέτη της οποίας την παρουσίαση ακούσαμε ακουγόταν μάλλον θετική ενώ υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά. Ή, είτε το θέλουμε είτε όχι απέτυχαν κάποια ε, ε, ε, επί της ουσίας απέτυχαν ορισμένα πράγματα ήταν η τύχη και μόνο τύχη το αν ε, ορισμένα πράγματα από τα κράτη-μέλη ε, είδαμε και είδαμε από το, ότι όταν αναθέτουμε πράγματα που γίνονταν πριν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα κράτη-μέλη τα πράγματα αποτυγχάνουν αυτό οφείλω να το πω Επίσης ήθελα να πω ότι οι περίφημες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν δεν είναι θέσεις ποιότητας. Τονίζω την ποιότητα εδώ. Και τελικά το, τα εισοδήματα θέλετε των οικογενειών ε, που πήραν για καινούρια θέση εργασία, δεν βελτιώθηκαν στην τελευταία ανάλυση. Ε, το επόμενο θέμα ε, που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στη μελέτη δεν αναφέρεται τίποτα και δεν αξιολογείται το γιατί δεν ε, γιατί η στρατηγική της Λισαβόνας δεν ήταν μια συνεπής πολιτική και μόνο βασιζόταν τελικά μόνο στα, στην τύχη και στις συμπτώσεις η επίτευξη των ορισμένων θετικών πραγμάτων. Η στρατηγική ε, της Λισαβόνας πρέπει να γίνει πραγματική στρατηγική. Αυτό πρέπει να πιέσουμε. Ε, Δημιουργηθεί ε, και τα λοιπά. Ίσως πρέπει να συζητήσουμε και τέτοια πράγματα, ξέρετε. Ο κύριος Τόμας Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ελίζαπεθ Σόντερ ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό. Ε, τι έγινε όταν ανέλαβα την εφαρμογή της Λισαβόνα στα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι πραγματικά μόνο τυχαίες συμπτώσεις οδήγησαν σε επιτυχίες. Είναι τρομερό αυτό. Πρέπει λοιπόν από εδώ και μπρο να προσέξουμε ποιες αρμοδιότητες μένουν στα χέρια των κρατών μελών και ποιες όχι σε τελευταία ανάλυση μπορεί οι διαδικασίες να είναι καλές ορισμένα πράγματα να εφαρμόστηκαν καλά αλλά ίσως δεν αρκούν γιατί χρειάζεται ε, να, ε, να υπάρχει περισσότερη συνεργασία και ενίσχυση των σχέσεων. Εγώ ρωτώ, σε τελευταία ανάλυση, αν αφήσουμε τα πάντα στα κράτη-μέλη που βρίσκεται η ευρωπαϊκή υπεραξία, αν θέλετε, η προστιθέμενη αξία πουθενά. Ε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε και να υποστηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πυρήνα και την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της στρατηγικής. Δεύτερο θέμα, κοινωνικό ταμείο. Το κοινωνικό ταμείο μπορεί να επενδύσει σε πράγματα στα οποία δεν μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση τελικά. Ε. Στον τομέα της εκπαίδευσης ε, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε επενδύσεις που να οδηγήσουν σε καλύτερη ποιότητα, όχι ποσότητα. Το, Ευρωπα... υπάρχει το ευρωπαϊκό σχέδιο ε, τίτλων, έτσι, qualifications framework. Ε, αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε να προχωρήσει, ε, να, τι να πω, συγκεκριμένα τώρα ρωτώ την Κομισιόν δεν μπορείτε να δείτε λεπτομερώς τι έγινε με τα εθνικά πλάνα, με τα εθνικά σχέδια δράσης, ποια από τα μέτρα των εθνικών ε, με κέντρων ε, σχεδίων δράσης, ποια μέτρα επέτυχαν αυτά να διαδοθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μάθει ο ένας από τον άλλον και να αναστρέψουμε κάποια στιγμή, αν θέλετε, τα πράγματα και να πούμε όχι ότι έχουμε κάποιους στόχους και εφαρμόζουμε μέτρα για τους στόχους, αλλά μάθαμε ορισμένα πράγματα τώρα. Από αυτά που μάθαμε δεν μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε σε στόχους για να δούμε μήπως πρέπει να αλλάξουμε τελικά στόχους. Άκουσα εδώ τώρα άλλους να μιλούν για τραγωδίες, άλλους να μιλούν για κομμωδίες. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή σκηνή, ωραία, αλλά εδώ δεν είναι παραμύθι η Ευρώπη. Είναι ο πολίτης που ζει και αυτό πρέπει να τον προσέξουμε. Δεν είναι θεωρη, θεωρητικό, θεατρικό έργο η Ευρώπη. Thanks very much. Um, <clears throat> well, we've Ευχαριστώ πολύ. Um, uh, Νομίζω ότι μου θυμίζει το έργο του Μπέκετ, περιμένοντας τον κοντό, όπου κάθονται οι άνθρωποι στη σκηνή και περιμένουν κάποιο, να συμβεί κάποιο υπερφυσικό γεγονός που θα λύσει για αυτούς όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς, εδώ και δέκα χρόνια, ο κοντό τον οποίον περιμένουμε δεν έχει ακόμα φτάσει ή αν έφτασε ε, δεν πρόλευε να μας ε, επηρεάσει. Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Δεν ε, Για την, για την ανάκτηση, για την ανάκτηση χρειάζεται ένα πιο μακροχρόνιο πλαίσιο για το οποίο θα χρειαστούν σοβαρές επενδύσεις απαιτεί να μην θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι θεός, αλλά να αντιλαθούμε ότι η αηφορία, η βιωσιμότητα σε, σε όλες τις διατάσεις, όχι μόνο την περιβαλλοντική αλλά και την οικονομική, την ε, ε, βιωσιμότητα της εκπαίδευσης ε, των πανεπιστημίων, των θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά πρέπει να εξαρτηθούν υπό το πρίσμα της αειοφορίας, όχι αποκλειστικά υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού. Οπωσδήποτε χρειάζεται και ο ανταγωνισμός, αλλά ομολογώ ότι με απογοήτευσαν οι Παρατηρήσει ε, του εκπροσώπου των επιχειρήσεων. Δεν άκουσα τίποτα το καινούριο από αυτά που έλεγαν πριν από 10 χρόνια σχετικά με τη στρατηγική. Η ευελιξία και η ασφάλεια δεν είναι επανάκια για την απασχόληση ή για να καταστεί ελκυστική η απασχόληση. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα από την ανεργία, από την ανεργία θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην απασχόληση πρέπει να είμαστε σοβαροί για αυτά που λέμε. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε το αδύνατο, να συντονίσουμε δηλαδή κράτη-μέλη την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική των κρατών μελών όταν μας, αποστερούν, μας στερούν το δικαίωμα να κάνουμε οτιδήποτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συμπράξουν και τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι αντιμετωπίζουμε μια βαθύτατη κρίση η οποία δεν θα ξεπεραστεί με τις παλιές λύσεις και τα παλιά μοντέλα. Βεβαίως πρέπει να έχουμε καλές υπηρεσίες υγείας, ε, ε, εκπαίδευση από την προσχολική μέχρι την ε, ηλικία, μέχρι την ανωτάτη εκπαίδευση. Οπωσδήποτε ευελιξία και ασφάλεια είναι κάτι το σημαντικό, αλλά με προβληματίζουν εκείνοι οι οποίοι δίνουν, δίνουν το βάρος μόνο στην ευελιξία δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να συνδυαστεί οπωσδήποτε η ευελιξία με την ασφάλεια, διότι αλλιώς θα οδηγηθούν στην απόγνωση οι άνθρωποι εάν το μόνο που λαμβάνεται υπόψη είναι η ευελιξία. πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία ανάμεσα εκείνους που προσφέρουν την εργασία και εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να αντλήσουν κέρδη από την εργασία. Η ποιότητα της επιτροπής που θα επιλέξουμε στο φέτος, η ηγεσία που θα αναλάβει αυτή την επιτροπή όλα αυτά τα οποία θα γίνουν ε, σε επίπεδο κρατών μελών, η ποιότητα του Κοινοβουλίου, ο ηγετικός ρόλος του Κοινοβουλίου, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. και κοιτάζοντας πίσω τα τελευταία δέκα χρόνια και να, και να λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ και κάτι άλλο εκεί, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Χρειάζονται πιο δυναμικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Ο κύριος Ίγκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι οποιοδήποτε λέει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας είναι μια επιτυχία, ασφαλώς ζει σε κάποιο διαφορετικό πλανήτη, όχι στον ίδιο πλανήτη στον οποίο ζούμε κι εμείς. Αν άκουσα σωστά, μια από τις επιτυχίες που αναφέρθηκε ήταν τα, βαλτικά, τα κράτη της Βαλτικής. Οι οικονομίε των κρατών της Βαλτικής ε, είναι σε άθλια κατάσταση. Η Λετωνία, η Λιθουανία και η Εστονία, οι, οι οικονομίες τους κατέρευσαν σημαντικά στο δεύτερο εξάμεινο του 2009. Η στρατηγική της Λισαβόνας έχει προωθεί ε, σαν κύριο, κύρια στρατηγική της ένα σκληρό ανταγωνισμό με θύματα τους εργαζόμενους και τις κοινωνίες. Η λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι μια πολυεθνική εταιρεία σαν την Dell να απολύει σε ένα κράτος μέλος πάνω από χίλιους εργαζόμενους και να μετεγκαθίσταται μετά σε ένα άλλο κράτος μέλος με τους εργαζόμενους που απολύθηκαν στην Ιρλανδία να εκπαιδεύουν ε, τους εργαζόμενους που τους αντικαταστήσουν. Η ΔΕ Επιτροπή να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να δωροδοκούν αυτή την πολυεθνική ώστε να φέρουν, φέρει αντιμετωπούς τους εργαζόμενους. Και οι Πολωνοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι όταν βολεύει την ΤΕΛ και βρούνε ε, εργατικό δυναμικό πιο φθηνό αλλού, θα εγκαταλείψουν ε, τους ε, Πολωνούς εργαζόμενους όπως εγκατέλειψαν και τους Ιρλανδούς. Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε για τραγωδία και κομμωδία αλλά μιλάμε για θέατρο του παραλόγου όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, πηγαίνει πριν από λίγες εβδομάδες ε, στην Ιρλανδία με 15 εκατομμύρια για ε, να προσφέρει ε, νέα κατάρτιση στους εργαζόμενους που είχε εγκαταλείψει η ΔΕΛ με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Η αιτία της κρίσης είναι ακριβώς η απελευθέρωση, η απορρίθμιση και η ιδιωτικοποίηση που είναι το λογικό αποτέλεσμα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Με άλλα λόγια, οι πολιτικές οι οποίες διέλυσαν τις οικονομίες του κόσμου. Στην Ευρώπη 29 εκατομμύρια άτομα είναι άνεργοι σε ένα χρόνο. Και τέλος κυρία Πρόεδρε, χωρίς κοινωνική ενσωμάτωση δεν υπάρχει τίποτα που να οδηγήσει κοινωνικό αποκλεισμό περισσότερο από ότι ανεργία. Και η στρατηγική της Λισαβόνα σημαίνει περισσότερη ανεργία. Δεν προσφέρει λύση στο θέμα. Επιτέλους το κίνημα των ε, ευρωπαϊκών συνδικάτων πρέπει να ξεπεράσει την προσήλωσή του στις αγορές και να αποφασίσει να εκπροσωπήσει δυναμικά τους εργαζόμενους από την Πολωνία μέχρι την Ιρλανδία για να αλλάξουμε αυτή τη στρατηγική αμφισβητώντας τη βάση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Σαρισαγιά και ο κύριος Κούπετς κατόπιν. arvoisa puheenjohtaja. Täällä puoluetaustasta riippumatta kuuluu... Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που, αυτό που έχει σημασία είναι τι νόημα έχουν αυτά τα συμβούλια και διαβούλια. Αυτό που ελέγχθη είναι ότι γίνονται πολλά βήματα ως προς το κείμενο, αλλά έγινε λόγος και για τα οικονομικά σχέδια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και φαίνεται ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία ευρία ανάλυση, έτσι ώστε οι μελλοντικοί μετασχηματισμοί να μας δώσουν καρπούς πώς θα αλλάξει η αγορά, η πράσινη αγορά και οι διάφοροι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί. Πώς η γύρανση του πληθυσμού θα έχει επιπτώσει στην αγορά εργασίας. Ποια, ποιες είναι οι απασχολήσεις, ποια είναι οι θέσεις μάλλον που θα εξαφανιστούν ο η συνάδελφος Γιάκον Σάρη, η Φιλανδή συνάδελφος, μίλησε για τις επιπτώσεις του ε, καλώς φέρεσθε και, τις, ε, αρμοδιο, και των και διαφόρων αρμοδιοτήτων ως προς τις γνώσεις. Η Κίνα ξεπερνά την ε, Ευρώπη στον τομέα του καλώς πράτην και της τεχνογνωσίας οι πολίτες αναμένουν από αυτή τη στρατηγική της Λισαβόνας την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εργαζομένων και την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων. Πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ε, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ως προς τους, ε, ως τις συνθήκες εργασίας που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πώς να αποφύγουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε σχέση με εκείνους που θέλουν να τηρήσουν τους όρους εργασίας των συλλογικών συμβάσεων. Εδώ χρειάζεται προστιθέμενη αξία της ε, συνθήκης ε, της Λισαβόνα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πουπάκης, η κυρία Έμιλι Τουρίνεν και έχουμε άλλη μία παρέμβαση. Και θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο ε, Ροντρίγκε. Ο καθένας μπορεί να ε, εκφραστεί ελεύθερα. Ο κύριος Πουπάκης. Από την περίληψη της μελέτης που άκουσα αλλά και από τους κοινωνικούς εταίρους θα ήθελα να επισημάνω ότι σε μια περίοδο που τα ποσοστά της ανεργίας είναι ιδιαίτερα αυξημένα και ένα μεγάλο μέλος, μέρος των συμπολιτών μας ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας εμφανίζεται μια ανησυχητική δυστοκία στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και κυρίως ποιοτικών θέσεων απασχόλησης με κίνδυνο η χρηματοπιστωτική κρίση να εξελιχθεί σε μια κοινωνική κρίση. Για να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη απορρίθμιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου απαιτείται η δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών τόσο στην κατάρτιση ενός νέου ευρωπαϊκού κοινωνικού προγράμματος όσο και στη διαμόρφωση των επιμέρους εθνικών σχεδίων σε κάθε χώρα. Πέρα δηλαδή από πρακτικές και πολιτικές που θα πρέπει να οριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να εκπονηθούν με κεντρική κατεύθυνση, ευρωπαϊκή κατεύθυνση, εθνικά σχέδια με ιδιαίτερη ακρίβεια και συνοχή και προγράμματα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να επιτευχθεί, αν θέλουμε, ο στόχο τη στρατηγική Λισαβόνα για καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα, την πλήρη απασχόληση, δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι ξαφνικά το παν η ευελιξία που οι επικεφαλής των επιχειρηματιών αυτή τη στιγμή φέρνουν εδώ μέσα και την κοινωνική συνοχή. Η κατάρτιση των παραπάνω σχεδίων θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες διαφάνειας, ευρείας διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής και της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σαν προϋπόθεση σε μια λογική τριημερίας με ισότιμη βάση, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο συνθήκες δημοκρατικότερης διακυβέρνησης. Η μέχρι τώρα συνδιαλλαγή σε εθνικό επίπεδο πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν έχει οργανωθεί σωστά με το αποτέλεσμα να μην εισακόγονται όλες οι απόψεις και ο κοινωνικός διάλογος, το λέω αυτό από πείρα γιατί συμμετέχω στις κοινωνικές οργανώσεις της χώρας μου, να μην γίνεται έγκαιρα και σωστά, να ξεφύγουμε επιτέλους από μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία σε κάθε χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται να επανεξεταστεί και να βελτιωθεί η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού στη βάση της ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, της άμβλησης των οικονομικών ανισοτήτων, τη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Έμιλη Τουρμένεν, και κατόπιν. Ε, ευχαριστώ. Θα πρέπει να μιλήσω αγγλικά δυστυχώς. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν για τα αποτελέσματα, για την έλλειψη αποτελεσμάτων και νομίζω ότι οι εργαζόμενοι της Ευρώπης εξακολουθούν να περιμένουν την κοινωνική Ευρώπη. Και αν ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που συνέβησαν το 2000, δεν υπάρχει βελτίωση. Αυξάνονται οι ανισότητες, εμφανίσετε κάτι που θεωρώ ότι είναι αμερικανική, ένα, μια, ένα αμερικανικό κόνσεπτ στο χώρο της εργασίας και σήμερα πλέον έχουμε κρίση με εκατομμύρια ανέργους. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να παραδεχθούμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση της Ευρώπης, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου, καθόλου καλή, κυρίως ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση και να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτον ότι αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να μείνει στα λόγια πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε τη, τη στρατηγική με την ε, διαμόρφωση, την ανάπτυξη της καλύτερης νομοθεσίας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ώστε να φέρει αποτελέσματα η στρατηγική της Λισαβόνας. Πρέπει να εμβαθύνουμε τη συζήτηση σε θέματα ουσίας πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αύξηση, ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, στην Ευρώπη, πώς θα δημιουργήσουμε την κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τους κοινωνικούς εταίρους, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό παράγοντας για την ανεπίδεξη των στόχων μας. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτε χωρίς αυτούς. Επίσης, στην Επιτροπή μας, και ελπίζω ότι κάποιος θα απαντήσει σήμερα σε αυτό, πώς θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουμε εμείς ως Επιτροπή ε, για τα πώς θα βάλουμε τα κοινωνικά και τα ζητήματα και τα θέματα της στο επίκεντρο, στο επίκεντρο αυτής της μελλοντικής στρατηγική. Θα ήταν σκόπιμο να το συζητήσουμε λίγο και αυτό. Θα σας απαντήσω σε ένα λεπτό για όλα αυτά τα σημεία. Η κυρία Ντανούτα Ζετλοβίκα θα είναι η επόμενη και τελευταία ομιλήτρια. Pan Rodriguez zwrócił uwagę na to, że strategia lizbońska nie była powiązana Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ροντρίγκες μας είπε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας δεν συνδέεται, συνδέεται πάρα πολύ λίγο με τον κοινοτικό προπολογισμό. Στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα μιλάμε για τις ε, οικονομικές προβλέψεις και προοπτικές πέρα από το 2014. Στο μέλλον θα είναι δυνατό να υπάρξει στενότερο σύνδεσμος ανάμεσα στα κοινοτικά κονδύλια και τη στρατηγική της Λισαβόνας δεν σκέφτομαι μόνο τα νέα κράτη-μέλη, αλλά όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ενισχυμένη δημοσιονομική σχέση θα μπορούσε να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους στόχους της στρατηγικής και θα ασκούσε και περισσότερη πίεση στις κυβερνήσεις που θα αισθανθούν ότι έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν στρατηγική. Κάτι άλλο. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα φόρουμ βέλτιστων πρακτικών για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Κάτι τέτοιο θα ήταν σκόπιμο να προωθηθεί θα ήταν μια καλή ιδέα αυτή για να προβάλλουμε τη στρατηγική, τη σε όλα τα κράτη-μέλη. Τέλος, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον τελευταίο μιλητή. Κυρία Τούρινεν, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να απαντήσουμε πώς θα συμμετάσχει η Επιτροπή μας σε αυτό το οποίο θα γίνει από εδώ και πέρα στη διαμόρφωση δηλαδή στρατηγικής 2000-2010 που είναι κάτι που θα χρειαστεί να, αναθεωρηθεί, να, να ανανεωθεί Ρίτσαρντ, μιλάω στην κυρία Τούρινεν, έχει σταθεί μπροστά και δεν τη βλέπω. Μου κρύβει την κυρία Τούρινεν. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το στάδιο δεν ξέρουμε ακόμα κάτω από ποιες συνθήκες συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλλει στη συνέχιση αυτής της διαδικασίας Εμεί η Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση και από εκεί και πέρα θα τη μελετήσουμε, θα διατυπώσουμε τις απόψεις ώστε το, την άνοιξη του 2010 να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Να εγκρίνουμε αυτό που θα αποτελέσει την επόμενη φάση. Πάντως να είστε βέβαιοι ότι εγώ, οι συντονιστές και τα μέλη του Προεδρείου θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ακουστεί η φωνή της Επιτροπής μας και να συμμετέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις διαδικασίες που θα αποφασιστούν, που θα περνάνε από τις Επιτροπές, τις ομάδες ή από κάποιες άλλες δομές. Σε τηλεγραφικό στυλ, επειδή φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης, ε, θέλω να δω μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει ή πρέπει να παραδεχθούμε ότι μεταξύ τραγωδίας και κομμωδίας δεν καταφέραμε να βρούμε μια απάντηση. και ε, επανερχόμαστε στην ανάγκη να κινητοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της θέσης του ε, σχετικά με τις ενιαίες, παραδείγματος χάρη, ε, κατευθυντήριες γραμμές. Πώς τι μπορεί λοιπόν να προτείνει αυτό το κοινοβούλιο ώστε η έξυπνη δουλειά που κάνουμε μαζί να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη. Τρίτο ερώτημα για την ευελιξία και την ασφάλεια. Νόμιζα ότι αυτή ήταν μια λέξη της μόδας πριν από ένα-ενάμιση χρόνο και ότι σήμερα λόγω της κρίσης στον τομέα της απασχόλησης που βιώνουμε έχουμε κάπως προχωρήσει πιο μακριά, πιο πέρα από την ευελιξία και ασφάλεια. Βεβαίως θα πρέπει να την προωθούμε και να την αναδεικνύουμε. Αλλά μήπως έχουμε φτάσει σε μια στιγμή που η πρόκληση είναι πώς θα διατηρήσουμε θέσεις απασχόλησης για να μην φεύγουν οι άνθρωποι από την αγορά εργασίας. Επειδή οι συνθήκες αυτής της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζουν αυτή την ευελιξία και ασφάλεια. Σε απαιτούμενο επίπεδο, ενώ αν βλέπουμε τα ποσοστά ανεργίας που έχουν φτάσει. Και ένα τελευταίο ερώτημα η δική μου εκτίμηση είναι ότι η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού ε, δεν ήταν αρκετά δυναμική. Η αναθεώρηση του 2005 επιδίνωσε τα πράγματα, διότι διατάραξε την ισορροπία της όλης διαδικασίας. Συμφωνείτε λοιπόν σε γενικές γραμμές με αυτή τη διαπίστωση ότι η αναθεώρηση του 2005 διατάραξε την ισορροπία και συνέβαλε και δεν επέτρεψε ε, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η σημερινή κατάσταση. Ακούσαμε 14 παρεμβάσεις στις οποίες θα σας ζητήσω να απαντήσετε σε ακριβώς πέντε λεπτά. Επιλέξτε τις, απαντήσεις, τις ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσετε. Ο κάθε ένας ε, βεβαίως έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στο, στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Και εσείς άλλωστε δεν έχετε καταλήξει, οπότε σας δίνω το λόγο για να συμβάλλετε και εσείς στη συζήτησή μας. Πραγματικά τα πέντε λεπτά δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Μπάς περιπτώσει, η ερώτηση του κύριου Θέρκας είναι πολύ δυσεπίλητη. Είναι πολύ δύσβατη ερώτηση, διότι ε, εμείς ε, είδαμε ότι υπήρξαν κράτη-μέλη τα οποία ήταν ενθουσιώδη ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές ε, στην παρακολούθηση των κατευθυντήριων γραμμών απασχόλησης και άλλα κράτη λιγότερο. Μπάση περιπτώσει, οι εθνικές ατζέντε υπερίσχυσαν. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ανάλογα με την ε, πολιτική απασχόληση, το κάθε κράτος μέλος έδρασε ε, προσπαθώντας να προσεγγίσει την ε, στρατηγική της Λισαβόνας. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο. Το 2005 μέχρι το 2005 ε, δίναμε ε, μεγαλύτερη, μεγαλύτερο βάρος στην απασχολησιμότητα και στην εφαρμογή των σχεδίων. Και αυτό ήταν ε, πολύ πιο εύκολο για 15 κράτη-μέλη. Μετά το 2005 αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ευελιξασφάλεια η οποία οδήγησε σε, μία, σε ορισμένες ανισορροπίες σε κράτη-μέλη και ε, υπερίσχεται ο σκέλος της ευελιξίας και όχι της ασφάλειας. Άρα οι επιπτώσεις αυτές, ε, αυτής της κρίσης ε, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές απασχολησιμότητας για το μέλλον. Έγινε λόγος για το θέμα της ποιότητα στην απασχόληση. Καθίσταται σαφές ότι το 2005-2007 δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο ποσοστό απασχόλησης, αλλά το 25% των ε, Ευρωπαίων εργαζόμενων έχουν ε, μισθό κάτω από 60% του εθνικού μισθού, δηλαδή είναι ε, φτωχοί εργαζόμενοι, όπως ορίστηκε εδώ αυτή η έννοια. Θα πρέπει να γίνουν πολλά ως προς τους μισθούς, το σύνολο των συνθήκων εργασίας και, εν πάση περιπτώσει, το σλόγγαν της ε, αναθεώρησης του 2005 ήταν πολύ καλό. Αλλά αυτό που είδαμε είναι ότι δεν κινηθήκαμε προς μία βελτίωση. Ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, λέχθη ότι τα κράτη-μέλη έδρασαν τυχαία. Όχι, είχαν μια εθνική ατζέντα και εφάρμοσαν την ατζέντα της Λισαβόνας. Μιλάμε για μια περίοδο 8-9 ε, ετών. Άρα, ορισμένα κράτη-μέλη μπόρεσαν να φτάσουν σε απτά ποσοτικά αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως υπήρχαν και άλλα στοιχεία τα οποία επηρέασαν περισσότερο από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Το ζήτημα όμως είναι πώς μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μία οδό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτό το name and shame δεν μπορεί να ισχύει παντού και πάντα, δηλαδή ε, κατονόμασε και στυλίτευσε. Αυτό, που έχει, αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να, να καταδείξουμε, να αποδείξουμε. Και για τη μελλοντική στρατηγική της ε, Λισαπόνας φαίνεται ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την τήρηση των υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη. Αυτό θα άρμοζε ιδιαίτερα, γιατί δεν θέλουμε ένα σύστημα naming and shaming, για εκείνους δηλαδή οι οποίοι δεν δέχονται αυτή την ε, βαθμολόγηση των κρατών μέλων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ποια ε, κράτη πληρούν τους όρους και σε ποια ε, χρονική περίοδο. Διότι αν έχουμε ένα, μια ιεράρχηση κοινών στόχων μετά το 2010. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε επακριβώς προθέσεις γιατί έχει μεγάλη σημασία από ποιο, ε, από ποιο ποσοστό ανεργίας ξεκινάει κανείς. Ως προς την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ε, καλή μέθοδος, αξίζει τον κόπο και μας οδηγεί σε μια μορφή συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Βεβαίως έχει ε, ελλείψεις, δεν υπάρχει πάντα διαφάνεια, τα ερωτηματολόγια που έχουμε συντάξει δεν είναι πάντα τα τα. Μερικά κράτη έμαθαν από άλλα, ενώ δεν ισχύει πολλές φορές το αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται ένα συντονισμός και ήταν ε, βεβαίως ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα. Η ευελίξ ασφάλεια μας δείχνει τι συμβαίνει στη, στην αγορά εργασίας διακρατικά. Έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και η ΟΚΕ έχει συντάξει μια έκθεση η, επ, της, ε, της έννοιας. Ίσως θα μπορέσει να μας ε, οδηγήσει στο να βγούμε από την ε, κρίση, αλλά αυτό μέσα σε λογικά πλαίσια. Έτσι ώστε να μην έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες. Για το 2010 και μετά θα πρέπει να έχουμε συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης από αυτόνομους οργανισμούς έτσι ώστε η αρχή της εύελιξης ασφάλειας να ισχύει σε όλες τις εθνικές αγορές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχατε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά αυτή είναι και η γοητεία αυτού του εγχειρήματο και, εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων η απόψινή. Μας είπατε ότι θα, μας, ε, θα είναι έτοιμη η μελέτη τον Οκτώβριο διότι όπως αντιλαμβάνεστε θα ήθελαν τα μέλη να έχουν την ευκαιρία να τη διαβάσουν το συντομότερο δυνατό. Κυκλοφόρησε ήδη ένα προσχέδιο, αλλά θέλουμε σε λογικές προθεσμίες να έχουμε ε, το πλήρες κείμενο της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει. Ερχόμαστε τώρα στην επόμενη μελέτη. για την οποία έγινε μια προσφορά πάντοτε στα πλαίσια αυτής της ευρύτερης συζήτησης ε, για τη συνέχεια που θα δοθεί στην στρατηγική της Λισαβόνας, αυτή ε, καλύπτει την συνεργασία ε, της, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η κυρία Τσέρα Καπαντή από το Ινστιτούτο το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών. Αυτή θα μας παρουσιάσει τη μελέτη και θα ακούσουμε κατόπιν εκπροσώπους ΜΚΟ οι οποίοι θα ε, κάνουν κάποια σχόλια. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Τεβαλή να μην ακολουθήσει το καλό παράδειγμα του προκατόχου σας και να τηρήσετε ακριβώς τα 15 λεπτά για να έχουμε περισσότερο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποια πρώτα στοιχεία για το θέμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μας ζητήθηκε να μελετήσουμε την εξέλιξη της ε, κοινωνικής ανοιχτής μεθόδου συντονισμού το, από το 2000 και δόθε, την ε, πανεπιστημιακή συζήτηση, ακαδημαϊκή συζήτηση που συνόδευσε αυτή την εξέλιξη το ρόλο και την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στην όλη διαδικασία, τη συνεργασία, την, ε, την αλληλεπίδραση OMC ε, της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία, το ρόλο των ενδιαφερομένων και η ε, πραγματικά ε, στα αποτελέσματα της μελέτης καταφέραμε να βάλουμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία και τις ευκαιρίες και τους, ε, τα, τους περιορισμούς αν θέλετε που υπάρχουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σχετικά με το θέμα αυτό. Ξεκινώ μιλώντας για το πώς η κοινωνική ανοιχτή μέθοδος συντονισμού συνδέεται με την ε, στρατηγική της Λισαβόνας. Στην ε, συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2000 έρχεται και οι κρατών και κυβερνήσεων ανέλαβαν τη δέσμευση να, ε, πήρε, να καταπολεμήσουν αν θέλετε τη φτώχεια μέχρι το 2010 και ζήτησαν από το Συμβούλιο να ορίσει, τους, ε, να ορίσει στόχους ε, οι οποίοι θα βοηθούσαν στον αγώνα αυτό και στην καταπολέμηση της του κοινωνικού αποκλεισμού. Είπανε δε ότι όλα αυτά θα βασίζονται στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και η από εκεί και πέρα πρόκειται να γίνει αναφορά, αν θέλετε, και αξιολόγηση όλων των ε, μέτρων και των διαβημάτων που θα γίνονταν κάθε χρόνο από κοινού, από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Μεταξύ 2003 και 2005 ε, ορίστηκαν οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ε, ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και εδώ καλύπτουμε ουσιαστικά, προσπαθούμε να καλύψουμε και την κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία και την, τις υπηρεσίες υγείας. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζήτησε ε, το ειδικά να προσέξουμε την κοινωνική ενσωμάτωση. Βεβαίως, όσον αφορά όλα αυτά τα, όλες αυτές τις πτυχές ε, συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μία οπτική γωνία θα ήταν να δούμε τις διαδικαστικές αλλαγές στη διαχείριση και στις διαδικασίες χάραξη πολιτικής. Άλλος τρόπος θα ήταν, άλλη οπτική γωνία θα ήταν να δούμε ε, ποιες αλλαγές κατά ε, κατά κύριο λόγο υπάρχουν τέτοιες διαφόρων ε, θεμάτων που καλύπτονται από τις εθνικές πολιτικές ατζέντε. Ε, τι κάνουν δηλαδή τα κράτη-μέλη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διαδικασίες για... και τη διαχείριση. Πολλά από τα μέτρα που πήραν τα κράτη-μέλη ε, έχουν ε, θετικά αν θέλετε αποτελέσματα τουλάχιστον φαίνονται θετικά ξεκινήσανε με ε, χάραξη ειδικών στρατηγικών σχεδίων δράσης κτλ και λόγω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού πολλές χώρες βελτιώνουν βελτίωσαν τουλάχιστον το συντονισμό των πολιτικών τους και σε το συντονισμό των πολιτικών σε διαφορετικούς τομείς, τα, το συντονισμό των επιπέδων διακυβέρνησης που εμπλέκονται και έτσι πολλά, βλέπουμε πολλούς αρκετή βελτίωση αν θέλετε και μέσω των δικτών που έχουν αποφασιστεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον από τα αποτελέσματα που έχουμε από τις διαδικασίες, από τη διαχείριση και τα λοιπά, βλέπουμε ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού είναι ένα καλό εργαλείο, το οποίο τελικά οδηγεί σε καλύτερο οριζόντιο συντονισμό και ε, ε, πολιτικές διατομεακές, αν μπορώ να το πω έτσι, και επίσης καλύτερο κάθετο ο, συντονισμό μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και σε ορισμένες περιπτώσεις τοπικών ε, κυβερνήσεων. Ε, ε, ενισχύεται αν θέλετε και προωθείται η συμμετοχή και μη κυβερνητικών βεβαίως φορέων και θεσμών αλλά υπάρχουν και αρνητικά σημεία ειδικά στο θέμα της άμεσης μάθησης, direct learning. Όπως είπα υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ε, διακυβέρνησης και στο θέμα της κοινωνικής ε, ενσωμάτωσης αλλά όχι παντού. Υπάρχει βέβαια το δυναμικό να έχουν παράγει θετικά αποτελέσματα και για τον τομέα της, μα... αλλά ε, εδώ τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν βεβαίως κάποια παραδείγματα direct άμεσης ε, μεταφοράς αν θέλετε πολιτικής από το ένα κράτος στο άλλο αλλά σε γενικές γραμμές δεν βλέπουμε να υπάρχουν ε, σημαντικά αποτελέσματα εδώ no ad Επίσης, ε, εκτός από το Progress δεν υπάρχει χρηματοδότηση έκτακτη που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαθέσουμε στην ε, υποστήριξη τέτοιου είδου μέτρων άμεσης μάθηση, όπω λέγαμε. Μπορεί και αυτό να παίζει κάποιο ρόλο. Απ' την άλλη μεριά, όμως, θετικά αποτελέσματα μπορούσε να δει κανεί ε, στην, ε, στις αλλαγές που έγιναν στην όλη φιλοσοφία που διέπει εθνικές πολιτικές. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαφνικά κάποιες ευρωπαϊκές έννοιες κατηγορίες ε, όπως το flexicurity, η ενεργή γύρανση, η ενεργή ενσωμάτωση κτλ. που είναι έννοιες ευρωπαϊκές, βλέπουμε ξαφνικά οι έννοιες αυτές να ενσωματώνονται στις εθνικές συζητήσεις ή, και ελπίζουμε μελλοντικά και στις εθνικές πολιτικές και έτσι ναι, οι, αυτοί που χαράζουν πολιτική στα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν μια καινούργια προσέγγιση, μια καινούρια φιλοσοφία, καινούριε ιδέες. Αυτό είναι καλό. Αλλαγέ τώρα σε εθνικές πολιτικέ και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων μα, θα μπορούσαν να ήταν περισσότερες, αλλά βλέπουμε να έχουν γίνει, να έχουν επιτευχθεί και αρκετές τέτοιες αλλαγές. Αλλά τουλάχιστον νέα θέματα τίθενται επιτάπητο στο ε, εσωτερικό επίπεδο των κρατών μελών και έτσι ε, ε, αυξάνονται και οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση νέων θεμάτων υιοθέτηση καινούριων προσεγγίσεων. Μια πρώτη αξιολόγηση αν θέλετε από, τα, από τις εμπειρίες που είχαμε με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού μας δείχνει ότι ε, ουσιαστικά η μέθοδος ε, δημιούργησε είχε θετικά αποτελέσματα, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν και αρνητικά σημεία. Μια ευρέως δεδομένη αντίληψη ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της φτώχειας και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή ε, ίσως είναι άδικη γιατί οφείλεται σε μεγάλο βαθμό όχι στην κακή πια αν θέλετε ανοιχτή μέθοδος συντονισμού αλλά και στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν νομοθετικά ή χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να καταπολεμήσουν ουσιαστικά τον κοινωνικό αποκλεισμό σε το χαμηλό τοπικό επίπεδο και την φτώχεια. Η, από εκεί και πέρα οι εθνικές πολιτικές δεν ε, περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της φτώχειας. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ ο, δεν φταίει η μέθοδος αν μπορούν τα πράγματα να βελτιωθούν τώρα από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να δούμε και ορισμένα άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν κατά την άποψή μου Ε, πράγματι η μέθοδος είναι καλή και ε, έχει δυνατότητες αλλά δεν εφαρμόστηκε ε, επαρκώς και σωστά στην, στις διάφορες πολιτικές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού συνήθως επικρίνεται γιατί θεωρείται ότι δεν είναι αρκετά δημοκρατική. Γιατί όντως δεν περιλαμβάνει θεσμικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγχρόνως δεν, η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων είναι αρκετά περιορισμένη στα περισσότερα κράτη-μέλη. Για την τελική έκθεση και αξιολόγηση θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον τυπικό, αν θέλετε, επίσημο ρόλο, που, τον πραγματικό ρόλο και τον ενδυνάμει ρόλο που θα μπορούσε να είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα βεβαίως, από νομικής απόψεως, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όντως θα είναι περιορισμένη και θα είναι τελείως συμβουλευτικός ο ρόλος ε, του Κοινοβουλίου. Όμως, ε, μάλλον αυτό θα έπρεπε να είναι από νομικές απόψεις. Αλλά τελικά στην πράξη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και κατά την τελευταία θητεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προσπάθησε να ενισχύσει το ρόλο του ε, ε, ε, ενισχύοντας αν θέλετε το ρόλο του στην κοινωνική προστασία, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στις υπηρεσίες υγείας και Και έτσι και υιοθέτησε πολλά ψηφίσματα ε, τα ε, που όλα τους υποστηρίζουν την ε, φιλοσοφία της ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης και συνεχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο ενεργή κοινοτική πολιτική που να χρησιμοποιεί το μέθοδος, ε, ανοιχτή μέθοδος συντονισμού. Στο μέλλον πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι όταν αν θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε και αναλύουμε αυτή τη στιγμή μέσα των εμπειρογνωμόνων μας το πώς κατάφερε το, το τι κατάφερε μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ανάλυση των επιτευγμάτων αυτών αν θέλετε θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Τώρα δεν έχω προτάσεις ε, τελειωτικές, έχω κάποιες προκαταρκτικές προτάσεις για τη βελτίωση της ε, ανοιχτής μεθόδου συντονισμού Ε, αυτή τη στιγμή οι πανεπιστημιακοί όπω σας είπα μελετούν, ε, ε ακαδημαϊκά μελετέ, μελετάτε η μέθοδος αυτή, ε, γίνεται μια κάποια ανάλυση και τελικά τα πρώτα συμπεράσματα λένε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον κάθετο συντονισμό και την αλληλεπίδραση επίδραση εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών ε, όπως επίσης και να πρέπει να ενισχύσουμε τον οριζόντιο συντονισμό μεταξύ ε, πολιτικών και να βελτιώσουμε τη συνεργασία και με άλλες επιτροπές και ομάδες υψηλού επίπεδου. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες, σε 15 λεπτά. Πιστεύουμε επίσης ότι η ενίσχυση της αμοιβαία μάθησης, αν θέλετε, θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να σημειώσουν τις βασικές, να διαπιστώσουν ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αν αυτές είναι κοινέ και έτσι θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να μάθουν τα μένα από τα δε. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η διάθεση και ενημέρωση για την ε, ανοιχτή μέθοδο συντονισμού να, και να ε, ενισχυθεί πρέπει να, να ενισχυθεί η πολιτική παρουσία, αν θέλετε, της ο, διαδικασίας αυτής. Ε, δημοσιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική για να δοθούν κάποια βασικά μηνύματα κλειδιά σε όλους για να ε, μπορέσουμε ε, να στηρίξουμε μετά και μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των όλων φορέων για την κοινωνική ενσωμάτωση. Κλείνοντας να πω ότι εκείνο που είναι σημαντικό είναι να ενισχυθεί και το πλαίσιο της ε, ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στον κοινωνικό τομέα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Θα πρέπει να ε, προς, γίνει προσπάθεια για ευρύτερες διαβουλεύσεις για ένα ζωντανό διάλογο, κοινωνικό διάλογο για παρακολούθηση αν θέλετε της εφαρμογής ε, των εθνικών μέτρων που αποφασίζονται. Ευχαριστώ. Ασφαλώς θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις, αλλά προηγουμένως θα ζητήσω τον Τζαν Τζονς, μέλλον της ε, Δικούς Επιτροπής ε, της Social Platform και ε, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής να μας μιλήσει για το θέμα της όχι παραπάνω από 7 λεπτά. Okay. Uh, very much. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να σας μιλήσω απόψε θα είχαμε φανταστεί ότι θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και στο προηγούμενο μέρος της συζήτησης, γι' αυτό θα δείξω λίγες διαφάνειες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για το κοινωνικό πλαίσιο χωρίς να αναφερθούμε στη στρατηγική της Λισαβόνας, διότι η αρχική στόχη της Λισαβόνας ήταν σαφώς η εξασφάλιση της ε, κοινωνικής ε, συνοχής και είχε προβλεφθεί ένα συγκεκριμένος πυλώνας για αυτό το σκοπό σε άμεση σύνδεση με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Από, μόλις ήρθα από τη Λουμπλιάνα όπου έγινε, έλαβε χώρα μια μεγάλη συνέντεση, συνάντηση με συμμετοχή ε, πάρα πολλών ευρωπαϊκών οργανώσεων η κοινωνική μας πλατφόρμα προωθεί την αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Αυτό που ήθελα να σας πω προηγουμένως, ότι έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία για το θέμα της στρατηγικής 2000-2010 σε συνεργασία με εργατικά σωματεία, κοινοβουλευτικέ ε, οργανώσει, κλπ. Ήρθαμε σε επαφή με τον πρόεδρο Νταρόσο και σημαντικού ε, αρμόδιου για τη λήψη αποφάσεων για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα αυτό που υπογραμμίζουμε, τη στρατηγική, δεν έχει φέρει αποτελέσματα, δεν έχει πετύχει τους στόχους της για τις οργανώσεις μας και οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε είναι σαφείς, η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη δεν συνέβαλε στην ε, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και γι' αυτό πιστεύουμε ότι έφτασε πλέον η στιγμή να αξιοποιήσουμε όλα τα θετικά στοιχεία που διαφαίνονται. Δεν θα μπορέσουμε, δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι λυπηρό αυτό, διότι έχουμε ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ πλήρες που καλύπτει έξι διαφορετικά κεφάλαια με 17 προτάσεις και πάνω από 100 διαφορετικές συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς μπορούμε να δώσουμε το προβάδισμα στους ανθρώπους και στον πλανήτη. Και αυτό το κάνουμε μέσα από τα διάφορα ε, κεφάλαια ώστε να έχουμε ένα αποτελεσματικό κοινωνικό μοντέλο πώς ε, να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε τα οικοσυστήματα, πώς ε, θα δημιουργήσουμε συμμετοχικές κοινωνίες, πώς θα προωθήσουμε ποιοτικέ θέσεις εργασίας, θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Ελπίζω ότι θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε όλα αυτά τα κεφάλαια γιατί αυτό θα βοηθήσει οπωσδήποτε στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Και τώρα έρχομαι στο κυρίως θέμα της παρουσίασης. Ακούσαμε σαφώς ότι ο συντονισμός ξεκίνησε με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης Υιοθετήθηκε το μοντέλο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού το 2000 με σαφή στόχο την εξάλληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Κάτι, ένας στόχος ωστόσο που δεν επιτεύχθηκε. Τα κύρια στοιχεία είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν το θέμα της καθορισμού κοινών στόχων. Είναι πρώτη φορά που πλέον υπάρχουν κοινοί στόχοι για όλα τα κράτη-μέλη ε, που είναι πρόσβαση σε δικαιώματα και σε υπηρεσίες, βελτίωση της διακυβέρνησης, συμμετοχή των ανθρώπων στη διαδικασία διακυβέρνησης για την απίτευξη των στόχων, των ξεκάθαρων στόχων που έχουν τεθεί για τα κράτη-μέλη. Για όσους από μας δουλεύουμε στην πράξη, υπάρχει δέσμευση για ένα ουσιαστικό σχέδιο δράσης. με σκοπό να εντοπιστούν τα προβλήματα, να εξεταστούν, να συζητηθούν με, τους, με τις ΜΚΟ την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εντοπίζουμε λοιπόν τα προβλήματα, καταρτίζουμε σχέδια και μετά παρακολουθούμε την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Μιλάμε δηλαδή για μια δυναμική διαδικασία που στηρίζεται σε κοινούς δείκτες με τους δείκτες αυτούς ε, μπορούμε να εντοπίσουμε τα σημεία ε, τους τομείς όπου ε, έχουν σημειωθεί επιτυχίες, εκείνους πάλι τους τομείς όπου χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις. Ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει στην πράξη και προσπαθούμε μέσα από κοινοτικές δράσεις και κοινοτικά προγράμματα να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και αυτές τις δυσκολίες. Στην, όλη, στην προσπάθεια αυτή εμπλέκονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και υπάρχουν επίσης προγράμματα ευαισθητοποίησης, μια πολύ δυναμική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο που λαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα υπόψη και προσπαθεί να τα αξιοποιήσει και να τα αναπτύξει. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί συνένεση, όπως υπογραμμίστηκε στη μελέτη. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια για να αντιληφθούν όλοι τις ε, πολλαπλές πτυχές, ε, τις φτώχες και να συμφωνήσουν σε κάποιους τομείς προτερότητας. Η φτώχεια ε, των παιδιών, των μεταναστών, Υπάρχουν δηλαδή ε, ορισμένοι τομείς όπου, που, στους οποίους απαιτείται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Τα, οι δείκτες, τα στοιχεία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Τα προβλήματα είναι σοβαρά, διότι δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία και δεν ευθύνεται και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε πολιτική βούληση στα πλαίσια της διαδικασίας της, Βαρκε... της ε, στρατηγικής της Πραγματική ουσιαστική βούληση να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό μόνο που ε, φαινόταν να προέχει είναι η δημιουργία θέσεων ε, απασχόλησης, αλλά όχι καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ε, επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Βεβαίως δεν υπάρχουν, διότι δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο στα κράτη-μέλη και σε, ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά σε, ό,τι αφορά τα, τις επιμέρους ανάγκες, αυτά που γίνονται δεν επαρκούν για την κάλυψη, για την ικανοποίησή τους. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικοί στόχοι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο και ουσιαστικό τμήμα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πολλές φορές η, όλη η διαδικασία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό γραφειοκρατίας. Στο Βέλγιο έχουμε όμως ε, και στην Ισπανία κάποια πολύ αποτελεσματικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί, αλλά δεν προβάλλονται επαρκώς. Εμείς ε, μπορεί που ασχολούμαστε άμεσα με το θέμα να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, αλλά το ευρύτερο κοινό δεν ξέρει τίποτα για τα προβλήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τι συμβαίνει με το θέμα της ανισότητας σε συνδυασμό με τη φτώχεια. Όλα αυτά ε, οφείλονται σε και προσπάθειες σε επίπεδο υλοποίησης. Και δεν υπάρχει διασύνδεση με το εθνικό επίπεδο, κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Τι γίνεται στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί το θέμα δεν συζητείται στα εθνικά κοινοβούλια και δεν προωθείται κατόπιν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο μικρές ομάδες ανθρώπων είναι πραγματικά, ε, έχουν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει και ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Έχουμε το, ετοιμάσει το κείμενο ε, για τη social platform που περιέχει μερικές σημαντικές συστάσεις μεγαλύτερη ε, προβολή των θεμάτων αυτών. Πρέπει να προβλεφθεί ένα συγκεκριμένος ρόλος για την ανοιχτή ε, και να προωθηθεί σημαντικά η χρήση, η εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού διότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η καλύτερη υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων. Απαιτείται κατακόρυφος και οριζόντιος συντονισμός με συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και ε, να εξασφαλίσουμε επίσης ότι θα εφαρμόζονται οι κατευθυντήρες γραμμές, διότι υπάρχουν ε, πολύ καλές κατευθυντήρες γραμμές που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Θα χρειαστεί λοιπόν μια μελέτη που θα αναλύσει τα θέματα της ε, αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων και μερών σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας. Επίσης, πρέπει να υπάρξουν στόχοι. Στόχοι για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ε, εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την ε, μέθοδο, ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για τα κοινωνικά ζητήματα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαδικασία της μάθησας. Η, κοινωνική, η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού για τα κοινωνικά θέματα πρέπει να λάβει τις αναγκαίες ενισχύσεις μέσω του κοινωνικού μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν οπωσδήποτε χρησιμοποιηθεί για την προσπάθεια εξάλληψης του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά αυτά τα οποία έγιναν δεν επαρκούν, γι' αυτό πρέπει να ε, εξασφαλιστεί ε, μεγαλύτερη ενίσχυση των διαφορετικών ταμείων και ότι οι κύριοι φορείς, η ΜΚΟ παραδείγματος χάρη, να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια αυτά, κάτι που δεν ισχύει, ότι υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα. Το Εμείς υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν νομίζω ότι έχει ωστόσο στη διάθεσή του όλα τα μέσα που χρειάζονται για να παρέμβει κάθε χρόνο. Θα θέλαμε να υπάρχουν εκθέσεις και συζητήσεις για την κοινωνική πρόοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με την δημοσίευση ενός πίνακα βαθμολόγησης της πρόοδου που θα σημειώνεται από χρόνο σε χρόνο. Και αυτά βεβαίως πρέπει κατόπιν να συνδεθούν με τις συζητήσεις που θα γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την αναθεώρηση της στρατηγικής κάθε χρόνο, μετά αφού κατόπιν, προτού φτάσουμε κατόπιν στη συζήτηση που θα γίνει σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει επίσης να δούμε πόσο πολύ είναι δεδεθμένη να προχωρήσει στον καθορισμό κοινωνικών προτύπων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, δεν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η αναγκαία πολιτική βούληση και εδώ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δικαίωμα σε αξιοπρεπή ζωή, σε σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν στο χαρτί, αλλά δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Κάτι θα δημοσιεύσει σε τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα δείχνει, που θα δείχνει ότι δεν έχουν καλυφθεί ορισμένα επίπεδα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα για να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι πραγματικά προσπαθεί η Ευρώπη να πετύχει τους κοινωνικούς στόχους που έχει θέσει προωθώντας ε, την, ε, τον, την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για τα κοινωνικά ζητήματα. Θα θέλαμε να υπάρξει δυνατότητα για όλες τις ε, κοινωνικές για όλες τις ΜΚΟ που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα να λάβουν μέρος σε μια ευρύτερη ε, συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έπρεπε να φύγω για ένα λεπτό αλλά νομίζω ότι όλα ελέγχθησαν εν τη απουσία μου. Η κυρία Λίσμπετ Λίν έχει το λόγο. Είναι η πρώτη γεγραμμένη. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Μας ε, εκπλήσει, μας σοκάρει όταν δούμε ποια είναι τα ευρήματα της ε, έκθεσης. Μιλήσαμε για τον συντονισμό στον ε, κοινωνικό τομέα, για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και όλες τις παρεπόμενες εργασίες και οι στατιστικές δεν ε, διοχετεύονται παντού στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη δεν μαθαίνουν από αυτό το μάθημα. Αυτό ακριβώς μας ε, κάνει να αγανακτήσουμε. Ε, περισσότερος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξαιρετική αυτή η ιδέα. Αν δείτε τι συμβαίνει επί τόπου στα κράτη-μέλη, πώς δέχονται τα εθνικά προγράμματα, δράσεις. Όλα αυτά τα θέματα είναι μείζονος σημασίας. Η στοχοθέτηση επίσης είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθεί η επίτευξή της. Μιλήσατε για την επικουρικότητα, υπ' αυτή την έννοια πρέπει να τηρήσουμε την επικουρικότητα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε όταν ορίσουμε αυτούς τους στόχους. Γιατί όταν μιλάμε για συντονισμό, μιλάμε για τη βέλτιστη δυνατή, είτε για τους ηλικιωμένου, είτε για τα άτομα με ανάγκες, όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, εάν δεν ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μία διαδικασία, τότε αυτή η διαδικασία, αυτές οι πληροφορίες κατασπαταλώνται. Θα πρέπει να υπάρξει και μια χρηματοδότηση. Η πρόοδος είναι πολύ καλή. Πολύ καλά τα διαρθρωτικά ταμεία χρειάζονται όμως μηχανισμοί χρηματοδότησης έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να επιτύχουν αυτά που καταφέρνουν οι άλλοι καλύτερα. Αυτή η ετήσια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Η πολιτική θέληση θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τουλάχιστον στα περισσότερα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι ορισμένα κράτη-μέλη επιτελούν ε, πολύ σημαντική εργασία, αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να μας απασχολήσει ως Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτή την πολιτική θέληση. Θα το αφήσω σε αυτό το σημείο, αλλά θα πρόκειται για μια συνεχή ε, συζήτηση και αναμένω και τις, την εξέλιξη τη, τη, του σκεπτικού. Κύριε Κρυπόλτη, μίλησε για το μέλλον. Για το μέλλον του Ευρωπαϊκού νομιού, κύριε Ακούτσα. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ για την παρουσίαση, η οποία ήταν αρκετά επικριτική, διότι μας έθεσε ενώπιον της πραγματικότητας και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, διότι εμείς ε, αισθανόμαστε την πίεση από τις εκλογικές μας περιφέρειες. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ε, αυτό το εκτιμούν όλοι ιδιαίτερα, δηλαδή την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης γνωρίζοντας ότι υποβαθμίζεται και πλήττεται από την κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε ακόμη περισσότερο σε θέματα κοινωνικής ε, συνοχής, διότι η οικονομική κρίση πλήττει την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα. Άρα φέρουμε ειδική ευθύνη για να δημιουργήσουμε αυτή την πολιτική ηγεσία υπήρχαν πολύ καλή, καλές συστάσεις, δηλαδή να συνδυάσουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, έτσι ώστε να τις ενισχύσουμε. Αυτό ακριβώς κάνουμε με το πρόγραμμα μικροπιστώσεων και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό μέσο για το μέλλον μας. Επίσης ε, είναι δική μας η ευθύνη να τονίσουμε αυτή την ε, πτυχή της ε, στρατηγικής μετά την Λισαβόνα. Δηλαδή όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, η ανθρώπινη δηλαδή διάσταση έχει μεγάλη σημασία και είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα ως προς την μεταστρατηγική της Λισαβόνας η επόμενη Προεδρία πρέπει να εργαστεί επί του θέματος και χρειάζεται η υποστήριξη του Κοινοβουλίου ως προς το ελάχιστο εισόδημα. Ξέρουμε ότι τίθεται σε κίνδυνο σε αρκετά κράτη-μέλη εξαιτία της ε, κρίσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας πίνα, πίνακας ε, ε, βαθμολόγησης. Ξέρετε ότι οι Ρωμά αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση εξαιτία των διακρίσεων και επειδή χάνουν και, τις θέσεις, χάνουν και την εργασία τους. Εμεί θα πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Αυτό εξαρτάται από εμάς και όχι από τους προσκεκλημένους μας. Αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω αυτούς που μας έκαναν τις δύο πολύ σημα... Ε, ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσει και ίσω ε, ίσως θα έπρεπε να καθίσουμε όλοι μας να αναρωτηθούμε τι θα γινόταν αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είχε παίξει σημαντικότερο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το ερώτημα βέβαια είναι θέλαμε να είχαμε τέτοιο ρόλο όταν πρωτομιλούσαμε για αυτή τη μέθοδο. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε επισκέψεις σε πολλά κράτη-μέλη και σε πολλά κοινοβούλια ε, και παλιότερα ε, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι ε, θέταμε την ερώτηση για το κατά πόσον συμμετέχουν τα κοινοβούλια στα ανοιχτή μέθοδο συντονισμού αν χρησιμοποιούν μάλλον το εργαλείο αυτό και μας κοίταζαν με απλανές βλέμμα στις περισσότερες περιπτώσεις Τώρα όμως που μάθαμε περισσότερα είναι πιο σημαντικό εφόσον είμαστε, ξέρουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει η μέθοδος αυτή, είναι πιο σημαντικό να το και εμεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πείσουμε είτε το Εθνικά Κοινοβούλια είτε την κυβέρνηση σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο ότι μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή και βεβαίω δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί διότι δεν είναι απλώς χρησιμοποιούμε τη μέθοδο και λέμε ωραία πράγματα αλλά πρέπει να υπάρχουν και απτά ε, να υπάρξουν και αυτά αποτελέσματα στο τέλος. Η ε, κοινωνική ενσωμάτωση. Ας ε, καθίσουμε λοιπόν να τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα μετά τη Λισαβόνα και η ιδέα ενός ευραίος βήματος, μιας αγοράς κατά την αρχαιολογική έκφραση όπου θα συζητιούνται όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Βεβαίως ε, υπάρχει και το άλλο θέμα του διαλόγου με τη συγκοινωνία των πολιτών και η διασύνδεση αυτών των δύο πραγμάτων. Νομίζω ότι πρέπει και αυτό να κάτσουμε να το σκεφτούμε και ίσως εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινωνική πλατφόρμα και τις συστάσεις που μας έδωσαν. Μια ιδέα είναι αυτή. Πρόεδρος, Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι ομιλητές στον κατάλογό μου. Ε, ίσως όμως θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με δυο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα να πω ότι στον τομέα αυτό υπήρχε μια κάποια αβεβαιότητα, δεν ήταν καθόλου σίγουρο το τι θα γίνει στον τομέα αυτό, αν θα πρόκειται για κομμωδία, για τραγωδία και τα για τραγέλαφο. Νομίζω ότι η ίδια η Κομισιόν βεβαίω θα φτιάξει τις προτάσεις της, αλλά εμείς κάπως ε, είπαμε, πήραμε μια θέση για το θέμα. Τώρα γιατί Γιατί όπως ελέγχθη μετά από 10 χρόνια Για να μην είμαι και πάρα πολύ σκληρή, βλέπουμε ένα φοβερό φλού εδώ. Και δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα με τη στρατηγική της Λισαβόνας λέγαμε και για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού λέγαμε τότε που τη φτιάχνουμε τη στρατηγική ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και να είναι πρώτη στη γνώση κλπ. κλπ, κλπ. Άκυρο αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Δε και δεν επιμένω να ξαναπούμε κάτι τέτοιο. Αλλά βλέποντα τα πράγματα πώς εξελίχθηκαν και η συζήτηση, έχοντας ακούσει και τη συζήτηση που έγινε εδώ, λέω Εν πάση περιπτώσει, εν πάλι να πω ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο έκανε την προεκλογική καμπάνια βασιζόμενο στη στρατηγική της Λισαβόνας και λέγοντας ότι ε, πρέπει κάτι να κάνουμε και τα λοιπά. Έκτοτε τα πράγματα άλλαξαν και μιλάμε τώρα για στρατηγική 2020. Ωραία. Moi, un objectif temps qui, a plus de lisibilité Εκείνο που θέλουμε πάντως, αν είναι δυνατόν, να θα ήταν να φτιάξουμε μια στρατηγική, η οποία να μην έχει βέβαια γεωγραφικές, ε, γεωγραφικούς απόϊχους, η στρατηγική της Λαφωσαβώνας δεν πειράζει, αλλά να έχει περισσότερη ουσία και να έχει και περισσότερες δυνατότητες να επιτύχει. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ε, είναι περίπλοκα, ε, πρέπει ναι, σίγουρα να κάνουμε κάτι. Μέχρι τώρα όντως τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ακούστηκε ότι θα πρέπει να γίνεται μια ετήσια συζήτηση. Μα αυτό το πράγμα υφίσταται ε. για θέματα απασχόλησης. Γίνεται ετησίως μια κάποια συζήτηση, διάλογος όπως θέλετε πείτε είναι πολύ σημαντικό βεβαίω να γίνονται αυτέ οι συζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια αν θέλουμε να μπούμε σε περισσότερο πρακτικά πράγματα, επιχειρησιακά μάλλον, ε, το, όντως θα πρέπει το Κοινοβούλιο να φροντίσει να ε, συντονίσει, να προωθήσει τέλο πάντων ένα συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ή κάποιε αλληλεπιδράσει μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που χρονίζουν στα χαρτοφυλάκια των διαφόρων επιτρόπων. Για μένα το πιο συγκεκριμένο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτό αυτά που θέλουμε να κάνουμε είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Τέλειο εργαλείο δεν είναι, ωστόσο είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει το Κοινοβούλιο για να βελτιωθούν τα πράγματα στον κοινωνικό τομέα. Τέλο πάντων, αυτά που έκανα μόλις τώρα είναι απλώ παρατηρήσεις. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Και μια και δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές στον κατάλογό μου, θα ήθελα... Α, συγγνώμη, ειδού, ειδού. Η κυρία Μπαστός και μετά η κυρία Κεπελντή. Mais pour réagir et pour euh, peut-être rebondir sur tel ou tel propos. Madame Bastos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο μετά από τις ε, παρατηρήσεις που έκανε η Πρόεδρος σε σχέση με την ε, στρατηγική της ε, Λισαβόνας, την οποία δεν πρέπει πλέον να αποκαλούμε έτσι, αλλά η Λισαβόνα είναι η πρωτεύουσα της χώρας μου. Όχι, σας διακόπτω δεν είπα. Ε, έχω το προνόμιο και μπορώ να παρεμβώ. Εγώ δεν είπα ότι εγκαταλείπουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που ίσχυε από το 2000 μέχρι το 2010. Μετά το 2010 θα μιλάμε για μεταστρατηγική της Λισαβόνας. Άρα ήταν ένα συμβολικό θέμα ορολογίας. Πίσω όμως από την ορολογία δεν είπα ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική, είναι μια συνολική στρατηγική, είναι το κατανόησα πλήρως. Είναι ένα θέμα συμβολισμού, ονομασίας. Και δεν σημαίνει ότι εξαλείφουμε τη στρατηγική. Παράλληλα όμως, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι αυτή η στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί ε, ένα ορόσημο όπου το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα ε, βρήκαν έναν ευρωπαϊκό χώρο ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης πέρα από τους άλλους πυλώνες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό νομίζω ότι η στρατηγική της Λισαβόνας με αυτή την ονομασία έχει έναν σαφή στόχο σε σχέση με την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για όλους τους φορείς που βρίσκονται ανά το κόσμο ως προς αυτό το ορόσημο, ορόσημο αποδοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν λάθος ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε όρους οι οποίοι ισχύουν γιατί βεβαίως ελπίζουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα λειτουργήσει πλήρως και θεσμικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε μια στρατηγική η οποία αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη και την στρατηγική σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το επιχείρημα ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Σοζέ Μανουέλ Ντοράου Μπαρόζο, είπε όχι στη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά στη στρατηγική του 2020, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να, να παρνηθούμε αυτό το, το ορόσημο το οποίο ήταν ύψης της σημασίας διαχρονικά και ορίζεται από την στρατηγική της Λισαβόνας και μόνον. Ξέρουμε ότι υπέστη τροποποιήσεις, ε, νέες εξισορροπήσεις, διότι είμαστε πολύ κάτω από τους απότερους στόχους, αλλά αυτό έχει σχέση και με περιπέτειες για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη τα κράτη-μέλη, ούτε οι κυβερνήσεις. Σχετίζεται με κυκλικά φαινόμενα, σύμφωνα με τους οικονομικούς κύκλους που γνωρίζουμε όλοι. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ε, αναφέρω αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να καταρρίψετε τη στρατηγική της Λισαβόνας, θέλετε να την κατονομάσετε διαφορετικά για να μην επέρχεται σύγχυση ως προς την ε, ονομασία αυτή. Ευχαριστώ η κυρία Καπάλτη. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να δίνω το λόγο κάθε τόσο σε κάποιον όταν ανακοίνωσε ότι έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Θα σας δώσω το λόγο επειδή έχουμε χρόνο, αλλά παρακαλώ να τηρούμε κάποια τάξη. Δεν θέλω να στενοχωρήσω, θέλω να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερο στη συζήτηση. Αλλά για να υπάρχει τάξη στη... και να τηρούμε τις διαδικασίες, ε, όταν θέλετε να ζητήσετε το λόγο, το ζητάτε έγκαιρα. Euh, Θα είμαι πολύ Σε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν ναι, έχουμε 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική ενσωμάτωση χωρίς να αναφερθούμε σε μακροοικονομικές πολιτικές που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν ε, και συνηγορούν υπέρ εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχεια, ανεργίας κτλ. πρέπει να λάβουν υπόψη τους λόγους, τι προωθεί τις στρατηγικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη κρίση στις ευρωπαϊκές οικονομίες από την εποχή της δεκαετίας του 30 με τεράστιες επιπτώσεις για την ευημερία απλών ανθρώπων. Και δυστυχώς ε, ε, όσο συνεχίζεται και γίνεται πιο σοβαρή η κρίση αυξάνεται και η φτώχεια. Γι' αυτό πρέπει διαρκώς να συνδέουμε τα προβλήματα από τα οποία υποφέρουν οι άνθρωποι με τη φτώχεια, την ανεργία και τις πολιτικές που προκαλούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Στην Ιρλανδία έχουμε 120 εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται για την κοκακόλα, που απεργούν για ένα μήνα τώρα επειδή αυτή η εταιρεία η οποία είναι μια από τις πιο κερδοφόρες στην Ευρώπη έφερε φώναξε 120 εργαζόμενους και τους είπε πρέπει να δεχτείτε μείωση κατά 50% του μισθού σας, γιατί πρέπει να αυξήσουμε την κερδοφορία μας. Α, μιλάμε για άντρες και γυναίκες, με μικρά παιδιά, με υποθήκες, με δάνεια. Και αυτές είναι οι φρικτές πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι όλο και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. εφόσον λοιπόν έχουμε μια οικονομική στρατηγική και μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια ηγεσία που δεν, δεν ασκεί πίεση και δεν παρεμβαίνει ε, για να εμποδίσει αυτές ε, τις πολυεθνικές εταιρείες να κάνουν αυτά που κάνουν, υποβιβάζει αντί να ανεβάζει το επίπεδο των εργαζόμενων στην Ευρώπη και όσο διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση θα, φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα το πρόβλημα και όχι μια λύση. I'm sorry, I will uh, talk uh, we work um, uh, Σχετικά με αυτή την έκθεση πάνω στην οποία έχουμε δουλέψει, αυτά που προέκυψαν από τη συζήτηση είναι πολύ σημαντικά, διότι πράγματι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με μεσοπρόθεσμα ε, για την αντιμετώπιση αυτές της κρίσης και της επιπτώσεις της σε θέματα φτώχειας, ανεργίας, έλλειψης πόρων σε ορισμένες χώρες για να εφαρμοστούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ε, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κλπ. Και οι προκλήσεις οι μεσοπρόθεσμες που είναι η γύρανση του πληθυσμού, η εισρωή μεταναστών, όλα αυτά τα θέματα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Όταν λοιπόν μιλάμε για ανάπτυξη ε, και οι οικονομολόγοι τα συζητούν αυτά, πώς ορίζουμε την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο η οικονομική ε, ευημερία, αλλά και κοινωνική ε, ανάπτυξη, κοινωνική ενσωμάτωση. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία τώρα, σήμερα, στο θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε έδινε το προβάδισμα σε αυτά τα θέματα στις συζητήσεις του με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και αυτό πρέπει να ισχύσει ακόμα περισσότερο από εδώ και πέρα, ώστε αυτή η μέθοδος να καταστεί ε, λιγότερο άτυπη και πιο αποτελεσματική στο να οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Και οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τις ΜΚΟ είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρέπει κάθε χρόνο να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο μια ευρεία συζήτηση για όλα τα θέματα με συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προβολή σε όλα αυτά τα θέματα, να ευαισθητοποιήσουμε του, η πολιτική ηγεσία στη σημασία της, ε, για το πόσο σημαντικό είναι να συμβαδίζει η οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ενσωμάτωση. δηλαδή με αυτή την κρίση είναι πλέον περισσότερο προφανής η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις μελέτες προσπαθώντας να καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι, το πρόβλημα της έλλειψης ε, πολιτικής βούλησης και πολιτικής ηγεσία είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει ως Κοινοβούλιο να ενεργήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ δεν λύσαμε κανένα από τα θέματα, αλλά κάναμε έναν απολογισμό και προσπαθήσαμε λίγο μαζί να συζητήσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Τελειώσαμε τις εργασίες μας, αύριο κατ' εξαίρεση η συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα είναι μια ε, συνεδρίαση συντονιστών και μόνο, που θα καθορίσουν τη στατηγική τις προτεραιότητες για τις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής μας. Σε, θα